Καλώς ορίσατε λοιπόν και πάλι αγαπητοί συνάδελφοι. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είπα της εκπροσώπου εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στην πρώην γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Εξ ονόματος της είπα της εκπροσώπου, ο Επίτροπος, ο κ.